Κοιτάξτε, έχει μεγάλη σημασία να ξεκινήσουμε αμέσως τη συνομιλία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Διευθυντή Κούν. AF, ε, PPI France, Γερμανική Ομοσπονδία Τραπεζών, τέσσερις συνομιλητές μας. καλωσορίζω τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, κύριο Αχτρή, που θα πάρει το λόγο αμέσως για να προχωρήσουμε μετά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ναι, ναι, θα πάμε κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ. Κύριε Κούν, είστε έτοιμος να αναλάβετε το λόγο. Έχετε πέντε λεπτά. <laughs> Λίγος χρόνος για 300 διαφάνειες περίπου. Έχετε το λόγο λοιπόν, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις θέσεις μας για, τους προτινόμενους, για τα προτινόμενα ρυθμιστικά μέτρα. Έχουμε μερικές διαφάνειες δεν ξέρω αν μπορούμε να τις προβάλλουμε σε κάποια οθόνη. Υπάρχει η δυνατότητα. Εντάξει, ας μην χάσουμε όμως χρόνο με όλα τα εισαγωγικά. Ε, ξέρουμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κτλ. Μπείτε στο ψητό. Καλώς, καλώς. Επομένως πάμε στην διαφάνεια περιθμών 4. Πολύ σύντομη εισαγωγή, όχι στην ε, ΕΤΕ, αλλά το είναι η υλοποίηση των εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού ή άλλων εντολών που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΤΕ λοιπόν έχει την ε, διαχείριση της υλοποίησης του μεγαλύτερου κομματιού του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και έχει και άλλες εντολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 35 εντολές, 40 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εγγυήσεις του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Άμεσα και έμεσα γίνεται αυτή η διαχείριση. Και στόχος μας είναι να έχουμε στο δυνατόν μεγαλύτερο πολλαπλησιαστικό μέγεθος και χαμηλό κόστος για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Πολύ σημαντικό είναι να αντιληφθούμε ότι αδίποτε αλλαγή στην νομοθεσία λόγω του μεγέθους των εντολών που διαχειριζόμαστε μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην υλοποίηση και γι' αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή και επιφυλακτικότητα εξετάζουμε κάθε πρόταση αλλαγής. Εν όλο, στην επόμενη διαφάνεια, όπως βλέπετε, είμαστε νομίζουμε ο φυσικός άμεσος εταίρος της υλοποίησης των, ευρωπαϊκών, των εγγύσεων από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό ή άλλων εντολών. Γιατί, γιατί είμαστε οργάνωση εγγεγραμμένη στη συνθήκη, έχουμε εγγεγραμμένο στο DNA μας, την υλο... στο DNA μας την υλοποίηση των στόχων των συνθήκων και βέβαια έχουμε ύψιστες προδιαγραφές για το δημοσιονομικό έλεγχο όπως προβλέπουν και οι συνθήκες και είμαστε η μόνη χρηματοπιστωτική οργάνωση του κόσμου που παρακολουθεί με το νίκη με το σίγμα τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προδιαγραφές και έχουμε κάθε δυνατότητα για εξασφάλιση απόλυτης λογοδοσίας στον προϋπολογισμό τον Ευρωπαϊκό. Άρα είμαστε ο φυσικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όντας όμως ταυτόχρονα και ακριβώς επειδή είμαστε το τέτοιο σπάνιο είδο και εφαρμόζουμε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, είμαστε φυσικό εταίρος και των κρατών μελών, των ε, περιφερειακών σωμάτων ε, ή φορέων για την υλοποίηση από κοινού ε, των πιο διαφορετικών χαρτοφυλακίων και επενδύσεων. Προτινόμενες τώρα βελτιώσεις για τον προϋπολογισμό. Λόγω αυτού του ιδιαίτερου και ειδικού ρόλου που έχουμε ως οργάνωση ευρωπαϊκή. Με ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στο εδάφιο 142 που αναγνωρίζει ρητά τη σημασία της ε, πραγματογνωμοσύνης μας και των δυνατοτήτων μας για υλοποίηση των, του έργου του Ευρωπαϊκού προπολογισμού, αλλά και την απλούστευση που προτείνεται στο νέο ε, ενώ σε σχέση με την εναρμόνιση των εκθέσεων και των προϋποθέσεων καταγραφής επιδόσεων, χωρίς παραπάνω βέβαια γραφειοκρατική επιβάρυνση. Προσπαθούμε να έχουμε στο δυνατόν πλήρη λόγοδοσία έναντι του νέου προπολογισμού. Δεύτερον, ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στις απλοποιημένες υποχρώσεις δημοσιοποίησης που αφορούν κυρίως τις μικρότερες επιχειρήσεις, όχι για τα μεγάλα έργα, αλλά τις μικρές επιχειρήσεις. Τρίτον, ευπρόσδεκτο θεωρούμε και το γεγονός ότι αν ένα δημοσιονομικό μέσο, χρηματοοικονομικό μέσο ευρωπαϊκό έχει ε, μετοχές μειονότητας, ε, μειονοψηφία σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θα υπάρχει ανάλογη εφαρμογή των κανόνων για τη δικαιώματα των, ε, της μειονότητας των ε, μετόχων. Επίσης, η σημαντική είναι η εναρμόνιση της ε, επεξεργασίας των επιστροφών και η διευκόλυνση των συνδυασμών έτσε ε, ε, και κοινωνικών ταμείων. Θα ήθελα ιδιαίτερα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για την επέκταση της πρωτοβουλίας μετά το 2017 για την ε, συνέχιση των εργασιών θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Επειδή ακριβώς η ΕΤΕ έχει τέτοια εμπειρία και ευρύ πεδίο δράσης ως προς τα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά μέσα και τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, έχει τεράστια σημασία να μην αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού την ώρα που ο αγώνας τρέχει. Και αυτό θέλουμε να το υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρηθεί η συνέχεια κάποιων κανόνων, τουλάχιστον μέχρι το τέλο τη. Τρέχουσα δημοσιονομική περίοδου, όπως άλλωστε αναφέρεται και στη νέα πρόταση. Και είμαστε ευτυχεί γι' αυτό. Επιπλέον θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι το, η Ευρωπαϊκή ε, εξωτερική εντολή της ΕΤΕΠ σε συνδυασμό με το ΕΦΣΕ που μπαίνουν μέσα στο πεδίο του νέου κανονισμού θα ισχύουν από το 2020 και μετά. Πράγμα το οποίο σημαίνει αλλαγές ως προς την υλοποίηση επιβραδύνοντας και ίσως και ενισχύοντας το κόστος. Γι' αυτό χαίρομαι που δεν επιβάλλεται εξ αρχής, αλλά μόνο μετά το 2020 αυτός ο συνδυασμός. Ιδιαίτερα θέλουμε να τονίσουμε ότι η ΕΤΕ έχει επιφυλάξεις στο αν θα πρέπει να εφαρμόζεται από τώρα, ενώ είναι υλοποιήσιμο μόνο μετά το 2020. Από την άλλη θα πρέπει να τηρούνται σε ένα νομοθέτημα όλοι οι κανόνες και αυτό πάλι διευκολύνει και εξασφαλίζει ασφάλεια ε, για να ολοκληρώσω το δυνατόν πιο σύντομα μια υγιής ε, διαχείριση κινδύνου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό είναι καθήκον των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των τραπεζών που έχουν τη δυνατότητα και να παρακολουθούν, έχουν τις ε, ε, δεξιό, έχουν την γνώση, τις ικανότητες να αξιολογήσουν κινδύνους και να αναλάβουν τα μέτρα όπως τα χρειάζονται. Ε, προς το παρόν σταματώ, περιμένοντας τις δικές σας ερωτήσεις. Έχουμε βεβαίως και παραδείγματα συνδυασμών της εντολής με το έτσε, ε, διαρθρωτικά ταμεία, επενδυτικά ταμεία και έτσι, αλλά δεν θα σας καθυστερήσω άλλο για να έχω τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα περνάμε στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, θα ήθελα να τονίσω κυρίως την δυνατότητα συνδυασμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Χρειάζομαι τις ε, διαφάνειες. Το νέο άρθρο 38.1 γ του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων και το ε, καινούριο άρθρο 39α ε, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα άρθρα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και γιατί το λέμε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι με τα νέα αυτά άρθρα η δυνατότητα συνδυασμού των ε, διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα προσφέρει μόχλευση και μεγαλύτερη προσθετικότητα στα κονδύλια των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε απορίες σας. Βλέπετε ότι σε ό,τι αφορά τα κονδύλια του των διαρθρωτικών και παιδικών ταμείων, η μόχλευση θα είναι μεγαλύτερη και άρα θα έχουμε ε, προστιθέμενη αξία στην πολιτική συνοχή. Και αν δείτε μόνο το πράσινο, βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη εφαρμογή, καλύτερη εκτέλεση και περισσότερη χρηματοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερη διαφάνεια παρακαλώ. Εδώ έχουμε τη, τις πρωτοβουλίες για τις μικρομεσαίες τράπεζες που έχουμε δρομολογήσει σε πολλές ε, χώρες μέλη. Θα επικεντρωθώ σε δύο παραδείγματα, αλλά έχουμε και άλλες περιπτώσεις της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Φιλανδίας και της Ιταλίας. Επίσης, ε, εγώ στάθηκα σε δύο παραδείγματα μιας μεγάλης χώρας όπως η Ισπανία και μιας μικρής όπως η Μάλτα. Στην Ισπανία για την περίοδο 2014-2020 ήδη έχουμε χρηματοδοτήσει 35.000 δάνεια περίπου. Ε, περίπου 33.000 ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν χάρη στην πρωτοβουλία αυτή. Και το ανέφερα αυτό ως καλό παράδειγμα συνδυασμού των κονδυλίων του Αναπτυξιακού Ταμείου και ε, περιφερειών της Ισπανίας που επίσης συμβάλλουν το 15 περιφερειών. Επίσης, έχουμε συνδυασμό του Τραμείου Στρατηγικών Επενδύσεων με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία που είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος ε, γιατί ε, έτσι εξασφαλίζουμε συμπληρωματικότητα και όχι ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης. Και έχουμε τη δυνατότητα να ε, έχουμε και την Εθνική Κεντρική Τράπεζα μαζί με την ε, ΕΤΕΠ ε, σε αυτή την πρωτοβουλία, κάτι που επίσης είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Καταλαβαίνω ότι επαναλαμβάνομαι, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είναι σημαντική η προστιθέμενη αξία και συμπληρωματικότητα στην πολιτική συνοχή χάρη σε αυτό το σχεδιασμό των διαρθρωτικών επενδυτικών ταμείων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ η κυρία από την μόνιμη αντιπροσωπεία των Γαλλικών Τραπεζών στις Βρυξέλλες. Euh, Καλημέρα σας. Από το γραφείο BPI France στις Βρυξέλλες. Θα παρακαλώ να περάσουμε αμέσω στην έκτη διαφάνεια γιατί δεν έχουμε χρόνο. Εισαγωγικά να σας πω ότι είναι η BPI France. Είναι η ε, Γαλλική ε, Δημόσια Τράπεζα Επενδύσεων με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε δανειοδότηση ε, των επιχειρήσεων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η Γαλλική Τράπεζα Επενδύσεων έχει μια ιδιαιτερότητα, εργάζεται με περιφερειακά γραφεία σε ένα περιφερειακό δίκτυο πάρα πολύ πυκνό. Γνωρίζουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά τις επιχειρήσεις κατά τόπους, τις ανάγκες της αγοράς εκάστοτε. Εδώ και 15 έτη και πλέον εμπλεκόμαστε στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων σε διάφορα επίπεδα, είτε πρόκειται για τα διαρθρωτικά ταμεία, ε, τα οποία διαχειριζόμαστε ε, για τις γαλλικές περιφέρειες, 150 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 και πρόκειται για χρηματοδοτικά μέσα κυρίως. Επίσης έχουμε και εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα λεγόμενης κεντρικής διαχείρισης ε, μέσω ε, του προγράμματος εγγύησεων που διαθέτουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, ε, να σας περιγράψω λίγο το πλαίσιο, αν μου επιτρέπετε, πριν περάσουμε στις προτάσεις μας. Η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων σήμερα και ιδιαίτερα των διορθωτικών κονδυλίων ε, αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις. Υπάρχουν δυσκολίες απορρόφησης των κονδυλίων αυτών, καθυστέρηση στην εκταμίευσή τους. Τα χρηματοδοτικά μέσα ε, έχουν δυσκολία να προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές, ιδιαίτερα λόγω της πολυπλοκότητας των κανόνων διαχείρισης των συγκεκριμένων ταμείων. Στα πλαίσια αυτών η αναθεώρηση του κανονισμού Omnibus καθώς και των κοινών διατάξεων που εφαρμόζονται στα διαρθρωτικά ταμεία είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτα. Δεν θα επανέλθω σε όλα τα θετικά του κανονισμού αυτού και της αναθεώρησης, απλώς να περιοριστώ ε, σε τέσσερα βασικά που θα θέλαμε να σας διαβιβάσουμε και θα θεωρούμε σημαντικά για την αναθεώρηση του κανονισμού έτσι ώστε να βελτιωθεί και να απλουστευτεί ακόμα περισσότερο η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Και ιδιαίτερα η λεγόμενη χρηματοπιστωτική μηχανική. Το πρώτο σημείο. Euh, Είναι να ενσωματωθούν οι ανακτόμενες ε, προκαταβολές στο δημοσιονομικό κανονισμό. Τι είναι αυτό. Σήμερα είναι ένα μέσο που χρησιμοποιούν διάφορα κράτη-μέλη για να στηρίξουν καινοτόμα έργα. Ε, στη βάση και στη φάση της έναρξης. Βασικά είναι ένα εργαλείο αυτό ε, επιμερισμού του κινδύνου που δεν ρυθμίζεται από πουθενά, από κανένα κανονισμό, ούτε των διευθυντικών ταμείων. Είναι όμως χρηματοδοτικά μέσα. Δηλαδή υπάρχει μία προκαταβολή που δίνεται στην επιχείρηση και η οποία σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης του έργου επιστρέφεται στο σύνολό της. Ε, και σε περίπτωση που δεν επιτύχει η προσπάθεια πάλι επιστρέφεται κατά αποκοπή ένα ποσό. Αυτή λοιπόν η ανακτώμενη προκαταβολή δεν αναφέρεται πουθενά σε κανένα κανονισμό και δεν μπορεί να κινητοποιείται υπέρ των καινοτόμων ε, επιχειρήσεων και αυτό είναι λυπηρό. Γιατί υπάρχει ένας κανονισμός για τις κρατικές ενισχύσεις στις καινοτόμες επιχειρήσεις και εκεί αναφέρεται ρητά αυτό το εργαλείο ως χρηματοδοτικό μέσο. Για να υπάρχει λοιπόν μια εναρμόνιση έτσι, κανονιστική, προτείνουμε να γίνει ρητή αναφορά ε, σε αυτές τις προκαταβολές στο δημοσιονομικό κανονισμό. Δανειζόμενοι τον ορισμό που ήδη υπάρχει ε, στον κανονισμό για τις κρατικές ενισχύσεις. Είναι ο Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία, αλλά και το, ο κανονισμός πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη. Δεύτερη πρόταση. Ενίσχυση ε, της ασφάλειας δικαίου των ε, χρηματοπιστωτικών ε, μεσαζόντων. Σήμερα υπάρχουν κάποιες διαχειριστικές αρχές που διαχειρίζονται ε, τα κονδύλια αυτά και αναθέτουν ένα τμήμα της διαχείρισης σε κάποιους τρίτους βεσάζοντες. Ε, Εδώ υπάρχει πρόβλημα ε, για την, στην ερμηνεία των κανόνων και των διατάξεων που ισχύουν λόγω περιπλοκότητας. Και αυτή η κατάσταση που επικρατεί δεν επιτρέπει την σωστή χρήση αυτών των κονδυλίων επιτόπου. Σας προτείνουμε λοιπόν αυτοί οι διάφοροι μεσολαβητές που μπορεί να είναι ευρω... εθνικές δημόσιες τράπεζες ε, επενδύσεων και έχουν δημόσια εντολή διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων να ε, μπορούν να θέτουν προς ε, αξιολόγηση ή ακόμα και προς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της διαδικασίας που ακολουθούν στη διαχείριση των κονδυλίων. Αυτό κάνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αναγνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα αρθρωτικά ταμεία. Και η ιδέα είναι να ε, δοθεί η ίδια δυνατότητα στις ε, δημόσιες τράπεζες επενδύσεων με την ΕΤΕΠ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Τρίτη πρόταση. Οι δύο προηγούμενες προτάσεις αφορούσαν το δημοσιονομικό κανονισμό και οι δύο επόμενες αφορούν ε, ουσιαστικά τα διαρθωτικά ε, ταμεία αυτά καθ' αυτά και τις κοινέ διατάξεις. Και πάλι εδώ πρόκειται για απλοποίηση των ε, κανόνων ε, δικαιολόγησης της χρήσης των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Στα πλαίσια των χρηματοδοτικών μέσων. Τι συμβαίνει εδώ. Υπάρχουν κάποια συστήματα χρηματοπιστωτικής μηχανικής που απαιτούν από το δικαιούχο τις τελικές ε, επιχειρήσεις ουσιαστικά ε, να επιστρέψουν κάποια κονδύλια. Στόχος είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να υπάρχει ένας έλεγχος μόνο εξάντε εκ των προτέρων επιλεξιμότητας του δικαιούχου και αυτή τη στιγμή εγκριθεί ο δικαιούχος και το έργο να μην γίνονται έλεγχοι στη συνέχεια. Απλώς να ε, συλλέγονται τα διάφορα παραστατικά και δικαιολογητικά. Κάναμε λοιπόν εδώ μία πρόταση τροποποίησης ε, αυτής της διάταξης που βλέπετε ε, στις οθόνες για να εξασφαλίσουμε την ε, διαχείριση κατά αυτόν τον τρόπο και να ελαφρύνουμε λίγο τις διαδικασίες. Θα υπάρχει πάντα έλεγχος βέβαια και πάρα πολύ εμπεριστατωμένος και εκ των υστέρων. Η τέταρτη πρόταση γίνεται αφορά στο άρθρο 38 που θα επιτρέψει στις διαχειριστικές αρχές να επιλέγουν άμεσα ε, δημόσιες τράπεζες επενδύσεων και με μεγάλη χαρά ε, είδαμε το άρθρο αυτό να ε, εντάσσεται στο συγκεκριμένο κανονισμό για τις διατάξεις Εδώ σας έχουμε παραθέσει την ε, εκδοχή που συζητάει το Συμβούλιο αυτό τον καιρό. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι σωστός ο κατάλογος ε, κριτηρίων με βάση το δίκαιο ανταγωνισμού. Στην πρώτη τελευταία παράγραφο που προτείνει το Συμβούλιο αναφέρεται ότι θα πρέπει κανείς να δικαιολογεί την ε, χρήση των διαθεωτικών πόρων ως προς τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι ενδιαφέρον ως επιχείρημα, αλλά αρκετά επικίνδυνο από νομική σκοπιά. Τι θα πει άμεση ή έμεση ωφέλεια. Θα θέλαμε να διαγραφεί η έμεση ωφέλεια. Γιατί είναι περίπλοκο και να δικαιολογηθεί και να αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Και ε, δημιουργεί ε, νομική αβεβαιότητα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε τι αναφέρεται αυτό. Ποια είναι η, η έμεση ωφελή, το έμεσο όφελος για τις δραστηριότητε αυτές. Και ένα τελευταίο για το άρθρο 38 για την άμεση επιλογή των δημοσίων τραπεζών επενδύσεων ε, να έχει αναδρομική ισχύ για να αποφευθούν διάφορα εμπόδια, θέσεω σε λειτουργία, σε ισχύ κτλ. Αυτή η μεταβατική περίοδος από τη στιγμή που συζητούμε τώρα μέχρι την ε, οριστική έγκριση του κειμένου. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Hardcore. Εκ μέρους Επιτροπής ο κύριος Μούσο. Schade. Dann, ähm, Κρίμα. Καλά. Για να δούμε. Οι συνάδελφοι τότε. Ο συνάδελφος Ashworth και η ταπεινότητά μου έχουμε μένει άναυδη, αλλά ας ακούσουμε πρώτα τον Ρίτσαρτ, αν τα καταφέρει. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ τους καλεσμένους μας για τις ε, ιδέες ε, που μας παρουσίασαν. Σημείωσα τις προτάσεις τους για την επιστρεπτέα προκαταβολή και άλλες διευκρινήσεις. Επίσης ασφάλεια δικαίου για, τις, για τους φορείς διαχείρισης. Συμφωνώ. Θα τα συμπεριλάβουμε αυτά στην έκθεση και επίσης ε, θα πρέπει να βρούμε μια πολύ δύσκολη ισορροπία ε, στον κανονισμό. Να άρουμε φραγμούς ε, ε, στην, είσοδο για να γίνει πιο φιλική προς το χρήστη, εξασφαλίζοντας όμως χρηστή διαχείριση και κατάλληλο έλεγχο. Τέσσερα σχόλια θα ήθελα να υποβάλω. Καταρχήν, συμφωνώ με τα σχόλια για τη σχέση μεταξύ των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των Ευρωβουλευτών έχει εκφέρει πολλές ανησυχίες ε, ως προς το θέμα αυτό. Πολλοί αντιλαμβάνονται τις συνέργειες που μπορεί να προκύψουν από την ε, διαχείριση, αλλά ε, υπάρχουν ανησυχίες. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η, ξεχωρισ... η διάκριση μεταξύ των δύο αυτών πηγών χρηματοδότησης και ω προ τη φύση του και ω προ το θέμα του κινδύνου που λαμβάνουν υπόψη. Ναι, μεν κάποια συνέργεια στη διαχείριση αντιλαμβανόμαστε, αλλά δι διαρωτώμεθα κατά πόσο αποτελεσματική θα είναι μια τέτοια ε, συνδιαχείριση λόγω των διαφορών μεταξύ των δύο ταμείων. επίση χρήση συνδυασμού το, της χρηματοδότησης. Κάτι τέτοιο υπονομεύει τις επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, ε, μας είπα συνάδελφοι. Και επίσης, ε, κάποια πιο γενικά θέματα. Πολλής λόγος έγινε για τις επιδόσεις, για, για ένα προϋπολογισμό που εστιάζεται στις επιδόσεις, που προσανατολίζεται στις επιδόσεις. Αυτό όμως ε, υπονοεί μία αντιπαράθεση. Καταρχήν, ε, το ζητούμενο κυρίως εδώ είναι η απλούστευση. Και απλούστευση για να μην ε, επιβαρύνουμε περαιτέρω τη διοίκηση, συμφωνώ. Αλλά υπάρχει και το θέμα ποσοστού σφάλματος της δήλωσης αξιοπιστίας του ΝΤΑΣ. Και εκεί δείχνει τον άμεσο τη σχέση αιτίου-αιτιατού μεταξύ της περιπλοκότητας της νομοθεσίας και του ποσοστού υψηλού ποσοστού σφάλματος. Επίσης, τι θα πούμε στους ψηφοφόρους μας, στους γεωργούς μας, στις τράπεζες, στις ΟΤΑ, στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλουμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα για τους δέκτες της χρηματοδότησης, για να μην έχουμε δαπανίσει όλο αυτό το χρόνο μόνο και μόνο για να καταλήξουμε σε μία έκθεση που είναι ε, εκτενέστερη και περιεκτική, αλλά πολύ λιγότερο απλή, πολύ πιο περίπλοκη δηλαδή, από την αρχική πρόταση. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αυτά ευχαριστώ τους καλεσμένους και α, τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και περιμένω και τις συμπληρωματικές τους παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Κιόρμαν, και εγώ ευχαριστώ τους ομιλητές μας. Ζητώντα συγγνώμη για την καθυστερημένη άφηξή μου. Έχασα τα πρώτα πέντε λεπτά. Και ίσως έχασα τον παράγοντα που θα συνέδε ίσως τα διάφορα στοιχεία των παρουσιάσεων για να καταλάβω καλύτερα τι πραγματικά μπορεί να επιτευχθεί με το ΕΤΣΕ και πού υπάρχουν τα σημεία όπου συναντά τις υποδομές και πώς μπορεί να λειτουργήσει ο παράγων μόχλευσης, ποιος τον υπολογίζει, πώς μπορεί να παρουσιαστεί αυτός ο παράγων μόχλευσης με συγκεκριμένα παραδείγματα και με κάθε σεβασμό προς τους ε, ομιλητές μας και την, ε, όλη αυτή η οργάνωση που είναι εξαιρετική. Θα ήθελα να επισημάνω ότι έχω ακούσει πολλά και αναφορές οι οποίες ε, φαίνεται να κινούνται σε ύψος 30.000 ποδών στη στρατόσφαιρστικά, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι συμβαίνει και τι συγκεκριμένα επιτεύγματα έχει φέρει όλη αυτή η υπόθεση. Μπορείτε να μας δώσετε λοιπόν παραδείγματα συγκεκριμένα του τι έχει προσφέρει το έτσι. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει μπορέσει κανείς να μας δώσει κάτι το πιστικό ότι εξυπηρετούνται οι στόχοι. Γιατί ακούγονται βέβαια οι στόχοι, η συμπληρωματικότητα και όλα αυτά δεν χρειάζεται να σας τα επαναλαμβάνω. Αλλά απτά τι έχουμε καταφέρει. Γιατί ξέρετε, δεν θα μου αρέσει καθόλου αν φτάσει η ώρα να αντιληφθούμε ότι κάναμε τόσα και τόσα και τελικά δεν επιτύχαμε τίποτα. Το να λέμε διαρκώ, γενικά ότι α, είναι πολύ ωραία, ότι η θεωρία μας λέει ότι θα τα καταφέρουμε και ότι όλα αυτά συμπληρωματικά μεταξύ του φέρουν αποτέλεσμα, δεν είναι ουσία. Θέλω να δούμε συγκεκριμένα αν έχουμε επιτύχει τους στόχους που είχαμε ορίσει. Ε, και επιπλέον δίνουμε και χρήμα, έτσι κύριε Κούλμαν. Κύριο Ρούμπιχ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση, γιατί βέβαια η οικονομία στην Ευρώπη χρειάζεται αυτή τη χρηματοδότηση και φυσικά στο θέμα του ποσοστού σφάλματος θα κριθεί και το αν πρόκειται για ε, εσκεμμένο σφάλμα, απάτη, αν υπάρχει κάποια άλλη παρατυπία λιγότερο σημαντική και όλα αυτά τα ζητήματα. Πού είναι αυτά δηλαδή τα λιγότερο ή περισσότερο τυπικά και σοβαρά σφάλματα που θα πρέπει στην ανάκτηση να ληφθούν υπόψη. Επίσης, θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι οι κίνδυνοι που βλέπουμε στη διαχείριση. Όταν έχουμε συμβούλους, παραδείγματι, στους οποίους οι αμοιβέ υπολογίζονται αναώρα, πώς γίνεται ο έλεγχος. Πώς υπολογίζεται ότι έχει δουλέψει τόσες ώρες ο σύμβουλος για να καταβληθούν οι σχετικές αμοιβέ. ή επιπλέον. Εάν διαπιστωθεί ότι πρέπει να ανακτηθούν χρήματα και πρέπει να γίνουν αγωγές γι' αυτό, δεν σημαίνει επιπλέον δαπάνη, επιπλέον κόστος. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε για το result-based budgeting. Τα έργα τα οποία χρηματοδοτούμε πρέπει να διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση ότι έχουν φέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα αμέσως, αλλά και ότι και σε 5-10 χρόνια αργότερα παραμένουν αποδοτικά σε σχέση με τους στόχους τους. Θα πρέπει λοιπόν να είναι όχι μόνο οικονομικά συμφέροντα, αλλά και νομικά γερά, στέρεα τα σχέδια τα οποία αναπτύσσουν. Δεν μπορούν να παραμείνουν μόνο στη θεωρία. Και το άλλο είναι ότι θα πρέπει η επιτήρηση των έργων να εξασφαλίζεται για να μην χάνονται τα κονδύλια με υψηλά ποσοστά σφάλματος που δεν μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Η Πρόεδρος. Έχω βάλει και το δικό μου όνομα στον κατάλογο των μιλητών και ως εισηγήτρια θέλω να πω μερικά πράγματα. Το πρώτο αφορά το πεδίο εφαρμογής. Υπάρχει ένα τμήμα που ισχύει από το 2020 και μετά. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε από τώρα. Δεν ξέρουμε τα προγράμματα για το 2020 και μετά, αλλά τη ρύθμιση θα την αποφασίσουμε από τώρα. Δεύτερη ερώτηση. Πρόκειται για χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία είναι διάσπαρτα σε διάφορα σημεία, δεν θυμάμαι σε ποιο κεφάλαιο, στο δεύτερο. Ε, ε, Ειδικέ διατάξεις, παράγραφος πρώτη τι αφορά τη σημερινή προγραμματική περίοδο. Γιατί μας μας έλεγαν ανέκαθεν ότι είναι κατεπήγον το θέμα. Γιατί τρέχουν προγράμματα και θέλουμε να τα επηρεάσουμε. Ε, ποια είναι αυτά και πόσα ε, είναι άμεσης ε, ε, εφαρμογής. Και μετά ποιος θα τα εφαρμόσει. Πολύ φιλόδοξα μας τα παρουσιάζεται. Και κύριε Σκούν έχει δίκιο ότι αν θέλουμε να παραλύσουν τώρα όλα θα πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες στη μέση των προγραμμάτων. Πού υπάρχει συγκεκριμένη αλλαγή και πότε. Και να ρωτήσω και την κυρία Μερβέη, ωραίο όνομα έχετε θαύμα, το αβασέρι Κιουπεράμπλα. Λέτε ότι δεν υπάρχει ορισμός για αυτή την προκαταβολή που είναι επιστεπτέα για να έχουμε και το νομοθετικό αποτύπωμα. Κύριε Μουσού, θέλετε να απαντήσετε εσείς και μετά πάλι εκπρόσωποι των τραπεζών. Δυστυχώς ε, η Γερμανική Δημόσια Τράπεζα ε, δεν ήρθε. Α, ζητώ συγγνώμη, ο πρόεδρος Αρτουή πρώτα. Ευχαριστώ. Εστερνίζομαι κι εγώ τα συγχαρητήρια που έδωσαν οι προλαλήσαντες, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι στόχος μας εδώ και ζητούμενο είναι η απλούστευση. Έχετε λοιπόν πραγματικές προτάσεις απλούστευσης. Θέλουμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή Ευρωπαϊκό Ταμείο Διαρθρωτικών ε, ε, Επενδύσεων. Δεν μπορούμε να απλουστεύσουμε ε, τα πράγματα, γιατί θα έχουμε και εμείς κάποιες ευθύνες όταν θα ψηφίσουμε τον κανονισμό. Και πολλές φορές ε, και εμείς ε, οι νομοθέτες ε, μπαίνουμε στον πειρασμό να υιοθετούμε περίπλοκες διατάξεις, γιατί πιστεύουμε ότι με τις λεπτομέρειες θα λύσουμε προβλήματα, αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο εύχριστο το αποτέλεσμα όσο το φανταζόμασταν. Και μερικές φορές έχουμε καλές προθέσεις, αλλά το αποτέλεσμα δεν μας δικαιώνει. Γι' αυτό και ίσως ε, θα πρέπει να είμαστε πιο επικριτικοί σε αυτή τη σωρία των κανόνων. Και προσοχή, γιατί όταν είμαστε κρατικές τράπεζες ή Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ε, μερικές φορές είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα και το σύστημα που μερικές φορές χρειαζόμαστε εμπειρογνώμονες ε, των οικονομικοτεχνικών για να βρούμε το δρόμο μας. Και πολλές φορές αυτές είναι οι επικρίσεις που ακούμε από τους ε, δικαιούχους που προσκρούν σε ένα ε, τείχο περιπλοκότητας. Θέλουμε πραγματικά μία πλούστευση. Γιατί θέλουμε το αποτέλεσμα της έκθεσης να επιφέρει απλούστευση, που όμως θα να φαίνεται και εμπράκτος, επιτόπου, όχι μόνο στα... στη θεωρία. Για να μην διαπιστωθεί χάσμα μεταξύ των αγαθών προθέσεων και των αναγγελιών και της ε, πραγματικότητας εμπράκτου εφαρμογής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε, σε αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση όπου νέα χρηματοδοτικά μέσα όπως σε δημοσιονομικές εγγύσεις, το έτσε και η πρόταση για την αηφόρο ανάπτυξη είναι χρηματοδοτικά μέσα που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον πρόεδρο ε, Γιουνκέρ μετά τη θέσπιση του ε, πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και, την, ε, και τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Και συμφώνησε για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους ε, το Κοινοβουλίο, αλλά πολλές υπηρεσίες και πολλοί φορείς χρειάστηκε να κοπιάσουν πολύ για να συνδυάσουν και να συναρμολογήσουν τους διάφορους κανόνες. Επίσης τώρα έχουμε το άρθρο 10 και το Omnibus που τροπολογεί τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, ε, ουσιαστικά αντλεί συμπεράσματα και διδάγματα από την πρώτη φάση εφαρμογής και υιοθετήσαμε μία προσέγγιση σε δύο στάδια. Καταρχήν, ε, δεν θέλουμε να παρεμποδίσουμε την ε, εύρυθμη εφαρμογή των προγραμμάτων του τρέχοντος πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου και αν κατάλαβα καλό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί καλωσόρισαν, χαιρέτησαν αυτέ τι αλλαγέ και θα πρέπει να να λάβουμε υπόψη κάποια διδάγματα για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και μην ξεχνάτε ότι ε, στους επόμενους μήνες θα εκπονήσουμε την πρότασή μας για το επόμενο μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και επίση θέλουμε ένα προβλέψιμο πλαίσιο, όπως προτείνεται στο άρθρο 10 για τα μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα της εγγύησης και το καθεξής. Έχουμε λοιπόν μια προσέγγιση σε δύο επίπεδα μία πρώτη φάση που προβλέπει ε, μία, κάποιες αλλαγές χωρίς την παρεμπόδιση των ε, εκκρεμών προγραμμάτων και στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα θέσουμε τα θεμέλια για ένα στιβαρό και πάγιο σταθερό πλαίσιο. Ευχαριστώ κύριο Σκούν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Βεβαίως ευχαριστώ για την ερώτηση για τη λειτουργία του ΕΤΣΕ και γιατί δεν υπήρχαν πιο πρακτικά παραδείγματα. Με 10 λεπτά χρόνο που μας είχατε διαθέσει, τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε παρά μια πολύ γενική και αφηρημένη παρουσίαση της νέας πρότασης. Αλλά παραδείγματα έχουμε πολλά και καθημερινά μπορούμε να προσφέρουμε για να εξηγήσουμε πώς εξασφαλίζεται ε, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του έτσι, ο μόχλευση δηλαδή, αλλά και άλλα συγκεκριμένα παραδείγματα και πολύ ευχαριστώ να σας τα υποβάλω. Μια άλλη ερώτηση. Πόσο κοστίζουν οι σύμβουλοι, πόσο κοστίζουν οι δικηγόροι. Πολύ σοβαρή και αξιόλογη ερώτηση. Προσπαθούμε το κόστος αυτό να το περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνατό. Γι' αυτό και έχουμε εσωτερική υπηρεσία νομική και όχι εξωτερικούς συμβούλους επιτοπλίστων. Τεχνικούς συμβούλους θα χρειάζεται, πάλι θα αξιοποιήσουμε τους δικούς μας μηχανικούς και τεχνικούς. Και αν κοιτάξουμε το κόστος των χρηματοοικονομικών μέσων και το επίτευγμα, είναι νομίζω μικρή αναλογία αυτής της επιβάρυνσης σε σχέση με το αποτέλεσμα. Αυτές νομίζω είναι δύο κύριες ερωτήσεις που με αφορούν. Και μια και δεν έχουμε χρόνο, θα αφήσω περιθώριο στους συναδέλφους από την BPI ε, να απαντήσουν στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι αν θεωρήσετε αυτή στόχο έχει κυρίως την εναρμόνιση των κανόνων διαχείρισης μεταξύ ε, χρηματοοικονομικού, δημοσιονομικού κανονισμού και λειτουργίας ε, των έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για δε την απλούστευση δεν θεωρούμε ότι είναι αρκετή. Και πιο πρακτικά προτείνουμε παρέμβαση σε δύο στάδια. Σε ένα πρώτο στάδιο υποβάλλουμε προτάσεις που θα έχουν ε, σαν αντικείμενο την αντιμετώπιση των πιο επιγόντων προβλημάτων, την αιτιολόγηση των δαπανών, ε, τη διευκρίνηση στο μέγιστο του τι εννοούμε αιτιολόγηση δαπανών και κινητοποίηση ε, για τα, για τα μέσα που κινητοποιούν οικονομικά μέσα και επίσης Προσπαθούμε να έχουμε στο δυνατόν πιο ενιαίες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου για τα ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να μην είναι και οι ε, συνομιλητές τους διαρκώς εκτεθειμένοι σε μια αβεβαιότητα που θα τους επέτρεπε να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά. Αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο ασφαλώς θα χρειαστεί εις βάθος ε, αναθεώρηση αυτού του ρυθμιστικού σώματος, του κόρπους αυτού που είναι και ο κανονισμός και όλα τα λοιπά, με ουσιώδεις αναθεωρήσεις και ε, προσδιορισμό των νομικών πτυχών, των ορισμούς και τα λοιπά, κατά τρόπο συγκεκριμένο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, στο πρώτο στάδιο η απλούστευση σημαίνει ο πρόεδρος Σας διακόπτω. Η ΜΠΕΠΕ, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει πάρει εντολή από τις περιφέρειες. Για διάθεση διαρθρωτικών ταμείων. Μου περιγράφεται μια από αυτές τις ε, εργασίες. Λοιπόν, τα Περιφερειακά Συμβούλια που είναι αρχή διαχείρισης στη Γαλλία μπορούν να μας αναθέσουν εντολή διαχείρισης διαρθρωτικών ταμείων, διαθεωτικών ε, κονδυλίων, τα οποία κινητοποιούνται μέσω των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουμε προσδιορίσει, με τις προτάσεις μας στις περιφέρειες, Φερρυπίν. Περιφερειακό Ταμείο Εγγύησεων, που στηρίζεται σε κονδύλια διαρθρωτικά, αφενός, και κονδύλια προερχόμενα από την περιφέρεια, τη χρηματοδότηση της περιφέρειας, αφετέρου. Οπότε θα μπορούσε ως τρίτο σκέλος να παρέμβει η ΜΠΕΗ, η γαλλική. Και η διαχείριση θα γίνει από την Γαλλίας σε επίπεδο περιφέρειας με συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της περιφέρειας. Και η Επιτροπή συνήθω περίπτωση τι απαιτεί ως δικαιολογητικά για να τύχετε τον, ε, της χρηματοδότηση από διαρθρωτικά ταμεία. Πολύ σύντομα να σας δώσω μια πρώτη απάντηση και στη συνέχεια η συνάδελφος Ελίρα Εγκουγέν που είναι ειδική θα συμπληρώσει. Πιο πολύ το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η, ερμηνεία των κειμένων. Δηλαδή καλούμαστε να συμμορφωθούμε στο σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται και προκαταβολικά σε σχέση με την διαδικασία επιλογής, επιλεξιμότητας, μέχρι το τέλος τη διαδικασία της υποβολής έκθεσης reporting στην αρχή διαχείρισης, την αποταμίευση, την εκταμίευση, την δικαιολόγηση των ε, ε, δαπανών και όλα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα στάδια για κάθε ένα από τα οποία πρέπει να τηρούμε τους όρους απόδειξης της δικής μας παρέμβασης με βάση την ερμηνεία όπως την εννοούμε εμείς, των ευρωπαϊκών διατάξεων. Και εκεί ακριβώς έχουμε το πρόβλημα, ότι αντιμετωπίζουμε πάντα πρόβλημα ως προς την ερμηνεία των διατάξεων. Και έτσι είναι πιο περιορισμένη η δική μας δυνατότητα παρέμβασης. Παράδειγμα, έλεγχη. Εθνική, Φερρυπίν για μια δράση που θα μπορούσε στο πλαίσιο της ίδιας νομοθεσίας πάντα σε μια περιοχή, σε μια ελεγκτική διαδικασία να κρυφθεί σκόπιμη, σε μια άλλη ελεγκτική διαδικασία από άλλο ελεγκτή, μη σκόπιμη. Άρα και θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση των κειμένων έτσι ώστε να διευκρινιστούν τα νομικά χαρακτηριστικά της διαχείρισης, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε και διάλογο με τις αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές ελέγχου σε εθνικό επίπεδο, για να απαντούνται τα ερωτηματικά μας, οι απορίες μας. Γιατί ποτέ κανείς δεν μας απαντά. Και οι δικηγόροι ακόμα έχουν πολύ διαφορετικές ερμηνείες. Δεν δεσμεύονται σε τίποτε και η Επιτροπή μας απαντά, Ευθύνη δική σας πώς θα το ερμηνεύσετε. Άρα δεν έχουμε πού να καταφύγουμε. Και αυτή είναι μια πρώτη απάντηση που μπορώ να δώσω για το τι θα πρέπει να προβλέψει η αναθεώρηση αυτή του κανονισμού καταρχάς και στη συνέχεια στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να υπάρχει λοιπόν μια εναρμόνιση της διαδικασία διαχείρισης εκ των προτέρων να μπορεί η Επιτροπή να μας πει «Ωραία, έχετε κάνει μια καλή επιλογή, είναι ασφαλής, είναι βέβαιη, μην ανησυχείτε, δεν κινδυνεύετε να βρεθείτε αντιμέτωποι με ε, μια ε, μη θετική διαπίστωση στο τέλος του έργου. Ο πρόεδρος, ε, ναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να καταπήρετε πολλά χαπάκια αγχολητικά με τόσο άγχος που έχετε. Αγχολητικά. Μα είναι, ναι, είναι όπως και το Conseil Juridique είναι Τι Λέει ο μιλήτρια. Oui, bonjour, Céline Σελίνα Γκυγέν, εργάζομαι και εγώ στην ΠΠΗ ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, και είναι πολύ λειτουργική η πρόταση αυτή γιατί περιορίζει πάρα πολύ το ΕΤΠΑ ε, στις επιχειρήσεις ε, το θέμα της ασφάλειας γιατί υπάρχει μια αιμορραγία χρημάτων για τους ελέγχους και υπάρχει πρόταση ακριβώς για να ξεκαθαρίσουμε πού σταματάει ο λογιστικός έλεγχος και πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα κονδύλια στο ΕΤΠΑ και στην παρακολούθηση ε, των αποτελεσμάτων των χρηματοδοτήσεων μας. Ο συνάδελφος Τσέλα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αυτά που ακούω τώρα μόλις. Και Υποθέτω ότι οι συνομιλήτριές μας είναι ε, εμπειρογνώμονες. Μας δείχνουν ότι ε, είμαστε σε μια καταστροφική πορεία και σε λίγο θα τρακάρουμε στον τοίχο. Και εγώ αμφισβητώ ότι είναι εμπειρογνώμονες. Ε, ε χώρες που έχουν πείρα, διοίκηση και ε, πάση κάποια τριβή με αυτά τα προγράμματα να έχουν τέτοια προβλήματα. Φανταστείτε τι συμβαίνει στις χώρες που δεν έχουν τέτοιες πρακτικές και τέτοιες εμπειρίες. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη η σύγχυση που ε, επικρατεί. Και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη συζήτηση για τους νέους κανονισμούς για να προχωρήσουμε σε μια σωστή λογική διαδικασία έτσι ώστε να πιάνουν τόπο το διορθωτικά ταμεία στην περιφέρεια εκεί που χρειάζονται. να δημιουργούν και απασχόληση και ανάπτυξη, να έχουν τη δυνατότητα να το πράττουν ενδιαφερόμενοι, να ενισχυθεί και να διατηρείται η ε, ανταγωνιστικότητα. Εδώ κινούμε από την υπόθεση ότι τα διαρθωτικά ταμεία μπορούν να συνδυαστούν με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό μου φαίνεται να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από ακόμα και αν είναι η επιθυμία των εμπνευστών αυτής της ιδέας. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή πώς θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τα ταμεία αυτά και να έχουμε και το απαραίτητο ε, προσωπικό ε, που να γνωρίζει και τα δύο θέματα τόσο καλά ώστε να μπορεί να τα συνδυάζει. Ένα λεπτό μόνο. Να ευχαριστήσω πριν λάβει το λόγο για να κλείσει ο κύριος Άσφορτ. Ξέρετε ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Εγώ θα επιθυμούσα να είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούμε σε μεγαλύτερο βάθος με το θέμα, πιο συστηματικά και να δούμε ε, και στην συνολική ε, εικόνα τι έχει νόημα με τις τροπολογίες, τι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, τι είναι άσκοπο και άστοχο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και ο συνάδελφος Ashworth θα πάρει το λόγο τελευταίο σε να κλείσει. Uh, <coughs> ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας για τις ομιλίες που μας έκαναν. Βέβαια μας άφησαν με περισσότερες απορίες παρά με απαντήσεις και αυτή η αβεβαιότητα δείχνει πόσο δρόμο έχουμε μπροστά μας για το δημοσιονομικό κανονισμό. Και αμφιβάλλω να έχουμε αρκετό χρόνο για το τιτάνιο έργο που έχουμε μπροστά μας. Πάντως ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες για τα σχόλιά τους και όπως είπαν και οι συνάδελφοι σήμερα, αν οι εμπειρογνώμονες έχουν πρόβλημα με τον κανονισμό, που είναι πιο εξοικειωμένοι, ε, σίγουρα ε, ο βαθμός ε, εφαρμογής του κανονισμού στα κράτη-μέλη θα απέχει πόρο από, από αυτό που επιθυμούμε. Και πραγματικά αρχίζουν και με ζώνουν τα φίδια για το κατά πόσο θα καταφέρουμε το σκοπό μας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και του διερμηνεί ε, για την υπέρβαση του ωραρίου. Λύεται η συνεδρία. Καλό σα απόγευμα.